Μπανέλ που αντικαθιστά ε, τον κύριο Χουάν Κάρλο Ζηράου Ταφιτάλ από τις 3 ε, Φεβρουαρίου 2016. Το Κοινοβούλιο σημειώνει ναι, την εκλογή της. Καλωσορίσατε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάδελφος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρει το δικαιωμάτιο.